θέλω να σας πω ότι τα πρακτικά της χθεσινής συνδρής Ολομέλειας ε, είναι διαθέσιμα. Αν υπάρχουν ε, παρατήσεις για τα πρακτικά ε, που δεν υπάρχουν, άρα δεν έχουμε να